Λοιπόν, συνεχίζεται η συνεδρίαση της Ολομέλειας. Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης και τα κείμενα που εγκρίθηκαν είναι διαθέσιμα. Υπάρχουν αντιρρήσεις για τα πρακτικά.